τελευταίος ο εισηγητή, Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο ε, σημείο τη ημερησία διάταξη, δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την καταπολέμηση της επιδημίας διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση αυτή συνοδεύεται από τον κύριο Νικολάη, εξ ε, ε, Βάμε Νικολάη της Ευρωπαϊκής Συμβουλίου και τον κύριο Πίμπαλξ, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο λόγο έχει το Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, Είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έλαβε την πρωτοβουλία αυτή να διοργανώσει την παρούσα συζήτηση και να επισύρει την προσοχή σε αυτό το σημαντικό θέμα. Θα ήθελα σήμερα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τους συμπροέδρους την κυρία Κρίστελ ε, Σαντεμόζε, την κυρία Λάτφορτ, τη Μαρίσα Ματίας και τον κύριο Μπουσουτήλ για ε, την ηγετική του θέση και την ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου για το Διαβήτη που κίνησε το ψήφισμα. Συνεχίζουν ε, να εργάζονται ε, ακούραστα για να αυξηθεί η επίγνωση της κατάστασης ε, και των προβλημάτων που προκαλεί στην υγεία ο διαβήτης. Τα χρόνια νοσήματα γενικά στην Ένωση επιβαρύνουν σημαντικά και τους ασθενείς και το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Αυτό απαιτεί μια νέα προσέγγιση συντονισμένη και αυξημένη συνεργασία. Η βασική λοιπόν πρόκληση εδώ σε αυτό το πλαίσιο απορρέει από το γεγονός ότι ζούμε περισσότερο αλλά δεν ζούμε αρκετά υγιεινά. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αναπτύσσουν διαβήτη και άλλα χρόνια νοσήματα. Οι επιπτώσεις είναι προφανείς. Αυξάνεται η πίεση στην υγεία μας και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ε, μπαίνουν στην αγορά εργασίας λιγότεροι νέοι για να πληρώνουν ε, αυξανόμενο δημόσιο κόστος. Και ο διαβήτης είναι όντως ένα από τα τέσσερα πιο συχνά χρόνια νοσήματα. 30 εκατομμύρια περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαγνωσμένοι διαβητικοί. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί και να φτάσει τα 40 εκατομμύρια το 2030. 10% του προπολογισμού της δημόσιας υγείας των κρατών μελών αφιερώνεται στην άμεση θεραπεία του διαβήτη και αντιστοιχεί σε 80 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς εδώ να υπολογίζεται το κόστος αντιμετώπισης των επιπλοκών ή των συγγενών νοσημάτων. Σήμερα ο διαβήτης ε, ούτε αντιστρέφεται ούτε θεραπεύεται. Οι ε, σημερινές θεραπείες δεν προλαμβάνουν την εμφάνιση της νόσου, ε, ούτε μπορούν να εξαλείψουν την απειλή των μακροχρόνιων επιπλοκών. Γι' αυτό θα πρέπει η των συγγενων νοσηματων σημερα ο διαβητης ουτε αντιστρεφεται ουτε θεραπευεται οι σημερινες θεραπειες δεν προλαμβανουν την εμφανιση της νοσου ουτε μπορουν να εξαλειψουν την απειλη των μακροχρονιων επιπλοκων γι αυτο θα πρεπει χρονια ε, ε, αντιμετώπιση να αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική διαχείριση, την εκπαίδευση και την έρευνα. Η πρόληψη μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο διαβήτης τύπου 2 που αντιπροσωπεύει 85 με 90% του συνολικού διαβήτη, μπορεί να προληφθεί με βασικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης υγιεινής διατροφής και της τακτικής σωματικής άσκησης. Τι μπορεί να γίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Τα ζητήματα υγείας είναι κυρίως και ουσιαστικά ε, υπόθεση των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αδρανούμε. Το Δεκέμβριο του 2010 το Συμβούλιο ξεκίνησε μια διαδικασία προβληματισμού σε σχέση με τα χρόνια νοσήματα και κάλεσε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσουν δράσεις για να βελτιωθεί η απάντηση στα χρόνια νοσήματα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η διαδικασία έγινε σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και κατέληξε σε ένα έγγραφο προβληματισμού. Γίνεται λοιπόν ε, σε υψηλό επίπεδο αυτή η ε, διαβούλευση και αναμένεται στο Συμβούλιο να ολοκληρωθεί του χρόνου. Η Δανική Προεδρία υποστηρίζει πλήρω αυτή τη διαδικασία και θα ε, χρησιμοποιήσει το εξάμεινό τη για να το προωθήσει όσο γίνεται περισσότερο αυτό το θέμα. Τα χρόνια νοσήματα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας στον τομέα της υγείας θα είναι στην ημερήσια διάταξη του Ατύπου Συμβουλίου Υπουργών Υγείας τον Απρίλιο στη Δανία, όπου θα συζητηθεί το θέμα της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης και δράσης των ασθενών. Αυτό είναι και ένα θέμα ε, διάσκεψης που θα διοργανώσει η Δανική Προεδρία στις 11 και 12 Απριλίου στην Κοπενχάγη. Χαίρομαι επίσης που έχω την ευκαιρία να ανακοινώσω ότι το φόρουμ για το διαβήτη θα ε, λάβει χώρα στις 25 και 26 Απριλίου. Συμπεριλαμβάνονται πολλοί ενεχόμενοι πολιτικοί, κυβερνητικοί, αξιωματούχοι, ε, επαγγελματίες υγείας, επιχειρηματίες, ε, ασθενείς θα εκπροσωπούνται σε αυτό το φόρουμ και η Ιθανική Προεδρία είναι περήφανη που έχει τη δυνατότητα να το υποστηρίξει. Η ε, Προεδρία είναι πεπισμένη ότι οι εκδηλώσεις αυτές όχι μόνο θα συγκεντρώσουν εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς, αλλά θα υποστηρίξουν και τη διαδικασία προβληματισμού για τα χρόνια νοσήματα που είναι καθοδόν στο Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Επίτροπε, γίνονται σημαντικέ προσπάθειε για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει των χρονίων νοσημάτων σε και του διαβήτη οι ε, εργασίες στο Συμβούλιο είναι ε, ένας μόνο κλάδος των προσπαθειών που συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαν και πρέπει να γίνουν περισσότερα όμως. Η σημερινή συζήτηση και το ψήφισμα που θα ακολουθήσει αύριο θα ε, βοηθήσουν να αυξηθεί η επίγνωση και η συνειδητοποίηση της πρόκλησης αυτής για την υγεία όλων μας. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας για το θέμα αυτό για να αναφέρω συνέχεια στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Ο Επίτροπος Πίβαλς έχει το λόγο. Πρόεδρε, βουλευτές, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη δέσμευσή του να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα όσων πάσχουν από διαβήτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τη μερίμνά σα. Δημιουργεί μεγάλο πόνο σε 32 εκατομμύρια Ευρωπαίου και τι οικογένειέ του ο διαβήτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του προβλήματος αυτού της επιδημίας αυτής. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε πλήρως την έκκλησή σας προς τα κατημέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για το σωστό διατολόγιο και την σωματική άσκηση, προκειμένου να καταπολεμηθεί και να προληφθεί ο διαβήτης τύπου 2, όπως εκφράζει και το ψηφισμά σας. Εδώ δεν μπορούμε να προλάβουμε όλες τις μορφές διαβήτη. Όμως, για τον διαβήτη του τύπου 2 γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά αίτια που τον προκαλούν η παχυσαρκία, η έλλειψη ε, φυσικής άσκησης, ε, γυμναστικής ε, και άσκησης, Αυτά είναι στοιχεία που επιβάρυναν την κατάστασή μα τα τελευταία 20 χρόνια. Περισσότερου από τους ε, μισού Ευρωπαίους έχουν τέτοια προβλήματα, όπω τα χεισαρκία. Ένα στα τέσσερα παιδιά από 6-9 ετών ήδη ε, είναι παχύσαρκα και έχουν πρόβλημα μέλλον πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2. Γι' αυτό η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ε, επικεντρωθεί στα αίτια που προκαλούν το διαβήτη την παχυσαρκία και την έλλειψη σωματικής άσκησης. Στο πλαίσιο αυτής της ε, σκέψης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 πρότεινε μια, μια στρατηγική για την ε, σωστή διατροφή και την σωματική άσκηση, προκειμένου να στηρίξει τις εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση του διαβήτη. Η στρατηγική ουσιαστικά στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των έμπειρων κατομελών ώστε να καθορίσουν κοινέ δράσεις και πρωτοβουλίες με ταξί νέων προσεγγίσεων για τη διατροφή όπως τα βασικά θρεπτικά συστατικά όπως πολλούνται στην αγορά τροφίμων των κατομελών. Έπειτα να κινητοποιήσουν τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να αναλάβουν δράση μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαιτολόγιο, την ε, σωματική άσκηση και την υγεία. Και βεβαίω εδώ να συμπεριληφθούν και όλε οι οργανώσει καταπολέμηση του διαβήτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εδώ ε, θα είναι τη δράση των μέσων μαζική ενημέρωση, των παραγωγών τροφίμων και των διαφημιστών προκειμένου να στηρίξουμε τα εμπορικά πρότυπα που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Τώρα κάποιες συγκεκριμένες δράσεις με παραδείγματα. Οι ερευνητικές πολιτικές της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπή. εδώ έχουμε συγχρηματοδοτήσει πολιτικέ και δράσει με 300 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον μέσω του έκτου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Στρατηγικέ που καταπολεμούν την παχυσαρκία, τον πραγματικό βάρο και τη διαβήτη. 7 ε, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν μόνο στο 2007 για την έρευνα σε σχέση με το διαβίτη και την παχυσαρκία. Και βεβαίω για όλα τα μεταδυτικά νοσήματα με ε, την ε, πρωτοβουλία μας υγιής διατροφή για υγιή ζωή ήδη κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια και κυρίως τονώσαμε την, ερευ... την έρευνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που αφορά τα προβλήματα και τα αίτια του διαβήτη. Ε, ήδη τα φρούτα και τα λαχανικά διανέμονται ετησίως σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα παιδιά μέσω του προγράμματος για τη σχολική διατροφή, μέσω μάλιστα των δράσεων για την εκπαίδευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις πρωτοβουλίες φυσικής δραστηριότητα, όπως με κατευθυντηρίες γραμμές για την φυσική άσκηση. Και βεβαίω στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει περιορισμό της ε, του βάρους που δίνεται στο μάρκετινγκ, στην ε, διαφήμιση των ε, ανθυγινών τροφίμων και στη στήριξη των υγιών τροφίμων για τα παιδιά. Εδώ λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε για την τόνωση της Εθνικής Υγειονομικής Περίθαλψης κατά του διαβήτη και τα εθνικά προγράμματα για την παρακολούθηση της επιδημίας του διαβήτη και το πόσο εξαπλώνεται. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ε, στο διαβήτη των νέων και των παιδιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την έρευνα και την υγεία μπορεί να συμβάλλει σε καινοτόμε λύσει στην αγωγή κατά του διαβήτη, την περίθαλψη των ασθενών και στο να καταλάβουμε καλύτερα πώ αλληλοσχετίζονται με άλλα νοσήματα ε, και άλλε παθήσει ο διαβήτη και τα αιτία του. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να δώσουν την απαραίτητη συνέχεια στην ε, Πανευρωπαϊκή Σύνοδο για τα μη μεταδοτικά νοσήματα. Και βεβαίως θέλουμε μια διαδικασία μελέτης και διαβούλευσης, περισυλλογής ε, σε συνδυασμό με τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους για να δούμε τι άλλες ευρωπαϊκές δράσεις μπορούμε να αναζητήσουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, βουλευτές ε, και οι εισηγητέ. Εδώ αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει επιδημία διαβήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε τα κατεμέρια στην προσπάθειά του να διαχειριστούν το πρόβλημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει προσεκτικά το ψηφισμά σα και το πώ να αναζητήσει ε, απαντήσει στην έκκληση συγκεκριμένα για περαιτέρω δράση. Συμφωνούμε με το Ευρωκοινοβούλιο ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερε προσπάθειε κατά του διαβήτη. Λόγου χάρη να προλάβουμε τον διαβήτη, ιδίω στην εξαπλωσή του μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, να στηρίξουμε του ασθενεί και να του χορηγήσουμε περίθαλψη ώστε να έχουν μια γεμάτη πλήρη ολοκληρωμένη ζωή. Και βεβαίω να έχουμε τα καλύτερα διαγνωστικά μέσα και τι δυνατότητε περίθαλψη ώστε να περιοριστούν οι ανεπιθύμητε παρενέργειε και οι περιττοί κίνδυνοι. Εδώ, όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει περισσότερη θέμενη ευρωπαϊκή αξία εάν αντιμετωπίσουμε τα αίτια των νοσημάτων αυτών τις κοινέ πηγές τους, όπως ε, ένα αίτιο που μπορεί να είναι παχυσαρκία ε, και όχι να βλέπουμε τα νοσήματα μεμονωμένα. Μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε από κοινού το διαβήτη μαζί με, άλλα, με άλλες χρόνιες νόσους. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει μια οριζόντια, σφαιρική προσέγγιση και όχι να υπάρχουν μεμονωμένες στατικές για μεμονωμένες παθήσεις. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει υπό το πνεύμα αυτό ότι έχετε απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει, να χαράξει και να υλοποιήσει μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά του διαβήτη και να αναπτύξει δράσεις στον τομέα αυτό. Τέλος, να σας βεβαιώσω ότι αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες κινδύνου που βάσει των ε, αποδείξεων που διαθέτουμε και των στατιστικών στοιχείων, από τι βάσει δεδομένων των κρατών εδώ θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε πλήρω το ρόλο μα στην καταπολέμηση παθήσεων όπω ο διαβήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ όλου. Θα ήθελα να σημειώσω στους εδώ παρισταμένους ότι στις 8 το βράδυ θα πρέπει να διακόψω την συνεδρίαση. Εάν δεν έχουμε ολοκληρώσει το θέμα αυτό και πάλι θα πρέπει να διακόψουμε στις 8. Και τώρα παρακαλώ τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να λάβουν το λόγο με τον κύριο Πουζουτήλ πρώτα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που συζητούμε το θέμα αυτό ε, σήμερα. Είναι δύο χρόνια που προσπαθούμε να οργανώσουμε τη σημερινή συζήτηση, να συζητήσουμε το ψήφισμα Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια μαζί με τους συναδέρφους μου που έχουμε εργαστεί για το θέμα αυτό. Τρία εκατομμύρια πολίτες επηρεάζονται στην καθημερινή του ζωή από το διαβήτη στην Ευρώπη και άλλα 2 εκατομμύρια που υποφέρουν από το διαβήτη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες δυσκολίες, πλέον δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ε, το 30% των διαβητικών δεν έχουν καν υπόψη τους ότι πάσουν από διαβήτη. Χωρίς να είμαι γιατρός γνωρίζω ότι έχουμε να κάνουμε ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα εδώ. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα συζητούμε το θέμα αυτό, το ζήτημα του διαβήτη. Οι ζωές εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης επηρεάζονται και θα πρέπει από κοινού να ε, κοινέ λύσεις. Πολλές φορές λέγεται ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Στην περίπτωση όμως του διαβήτη το επιχείρημα δεν ευσταθεί. Εάν μπορούσαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του διαβήτη θα ξεκονομούσαμε πάρα πολλά χρήματα θα μειώναμε σε μεγάλο βαθμό κόστος που θα, μας, που θα βρίσκαμε μπροστά μας αύριο. Και γι' αυτό θέλουμε η Ιδανική Προεδρία να στηρίξει τις προσπαθίες μας. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια στρατηγική για την καταπολέμηση του, στρατιού, του διαβήτη και τα κράτη-μέλη να προτείνουν εθνικές στρατηγικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάλτε Μόζε, δεύτερη για μισή λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Πρέπει να δράσουμε και αυτό σημαίνει πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα για το διαβήτη. 32 εκατομμύρια πολιτών της Ευρώπης πάσχουν από διαβίτη. Άλλα 32 εκατομμύρια θα νοσήσουν σύντομα. Οι μισοί από αυτού υποφέρουν από διαβέτη τύπου Β. Τύπου διαβέτη Β, ο οποίος μπορεί να προληφθεί. Και γι' αυτό χαίρομαι που ακούω ότι συμφώνεται ότι πρέπει να δράσουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε προληπτικά και να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που οδηγούν στο διαβήτη, την παχυσαρκία. Πρέπει να ε, δώσουμε κίνητρα στον πολίτη να ζει κατά τρόπο πιο, πιο υγιή. Πρέπει επίση να βελτιώσουμε τη συλλογή των δεδομένων για το διαβήτη και άλλους τύπους ε, ασθενειών. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Και να ξέρουμε αν προχωρούμε, εάν με την υιοθέτηση πολιτικών πρωτοβουλειών ε, επιτυγχάνουμε κάποια πρόοδο. Εγώ άκουσα μεγάλη χαρά το Συμβούλιο που είπε ότι σκοπεύει να επιληφθεί του θέματος. Αλλά τα κράτη-μέλη αυτό που θα πρέπει να κάνουν θα είναι να θέσουν ε, σε ισχύ ε, εθνικά προγράμματα δράση του διαβήτη, γιατί και σε εθνικό επίπεδο μπορεί κανεί να λάβει δράση. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που δεσμεύεστε να δράσετε για του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η Βαρόνι Λάτφορντ έχει σα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ορολογιακή βόμβα του διαβήτη έχει σταματήσει απλώ να τρέχει και έχει ήδη εκραγεί. Χαίρομαι λοιπόν που η Δανική Προεδρία, όπω και το Κοινοβούλιο, ε, ασχολούνται με το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο βεβαίω εδώ έχει και δανεικέ επιρροέ. Και ασχολούνται ακριβώ με το διαβήτη ω προτεραιότητα. Εδώ πρέπει να δούμε το κόστο και για το σύστημα υγεία μα, που είναι αρκετό λόγο να μα απασχολεί το θέμα αυτό. Ήδη η εξάπλωση του διαβήτη στο παιδιά και στου εφήβου και η διάγνωσή του ε, στον τύπο 1 είναι κάτι βέβαιο για τον τύπο 2 δεν ε, είναι τόσο βέβαια και βεβαίω πολλέ φορέ ταυτίζεται και με άλλε ασθένειε όπω οι καρδιακέ παθήσει, η, ε, η τυφλότητα και ούτω καθεξή. Ε, στοιχεία που έχουν μεγάλο κόστο για το σύστημα υγεία. 15% όπω είπα έχουν τον τύπο 1 του διαβήτη, ακόμη και νεογνά. Εδώ λοιπόν χρειάζεται προφανώ μια οριζόντια προσέγγιση σφαιρική που όμω για την ώρα δεν έχει λάβει υπόψη παρκώ τον τύπο 1 διαβίτη. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε τα εξή σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα πώ αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον διαβήτη. Ε, δεν ασχολούνται απαρκώ με την διατροφή του. Πιστεύουν ότι αν δεν πεθάνουν από αυτό που τρώνε ε, είναι αρκετό να το, δίνουν αρκετή προσοχή στο διατολόγιο τους. Επίσης, για τον τρόπο ζωή που ακολουθεί κανεί, δεν αντιλαμβάνεται πόσο λανθασμένο μπορεί να είναι σε σχέση με το διαβήτη και πόσο μπορεί να προκαλεί και να επιβαρύνει την πάθηση. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πραγματικά μια οριζοντία προσέγγιση. Η ανάπτυξη μια ε, στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βάσει των συστάσεων του Συμβουλίου. Αλλά όχι αυτή που μα έχει προτείνει ω τώρα, διότι μέχρι τώρα τα μέτρα που έχουν ε, ανελθεί αλληλαποκλείονται. Ευχαριστώ. Του πρασίνου τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπρέπολς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη σε ένα ψήφισμά του στις 15 Σεπτεμβρίου του 11 εν ώψη ε, της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για μη μεταδοτικά νοσήματα δήλωνε ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται πάρα πολύ και θα πρέπει να αντιμετωπίσει ε, οπωσδήποτε και μέσω των αρμοδίων αρχών στα κράτη-μέλη αυτό το θέμα. Είχαμε και μια κοινή συνεδρίαση διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2010 ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ομάδα εργασίας για το ε, διαβήτη, για την καρδιά της Ευρώπης κατά των καρκίνων και ε, άλλα και μια άλλη ομάδα εργασία που είμαι εγώ πρόεδρος. Η πρόληψη λοιπόν είναι εκ των όνων κάνευ και είναι και δυνατή. Γιατί οι παράγοντε κινδύνου για όλες αυτές τις ασθένειες είναι γνωστοί. Λυπάμαι λοιπόν λίγο που έχουμε αφήσει τη συνολική προσέγγιση και κάνουμε πια ειδικό ψήφισμα μόνο για το διαβήτη. Υπάρχει προστιθέμενη αξία στο περσινό ψήφισμα ε, και μου λείπει εδώ γιατί υπάρχουν και άλλα μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως είναι οι καρδιαγιακές παθήσεις, ε, οι αναπνευστικές παθήσεις, ο καρκίνος. Είναι λίγο στην άκρη, έχουν παραγωνιστεί. Δεν έχω πρόβλημα με την ουσία του ψηφίσματος, βεβαίως το υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Και η κυρία Ματίας, τελευταία εκπρόσωπος από τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ήδη ακούσουμε, ο διαβήτης επηρεάζει πάνω από 30 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη. Και ε, βεβαίω πλήττει ιδιαίτερα και την οικονομία. Έτσι, δικαιολογείται το να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να ετοιμάσουμε ψήφισμα για το θέμα αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι η πρώτη φορά που το Ευρωκοινοβούλιο απασχολείται με το θέμα αυτό. Μιλάμε για μια συλλογική εργασία ε, μια προσπάθεια που δεν ακυρώνει όσα έχουν γίνει ω τώρα ως προσπάθειε ίσα ίσα τι ενισχύει τι προηγούμενε προσπάθειε και τη δυνατότητα που διαθέτουμε να δρούμε από κοινού. 300 εκατομμύρια θανάτους έχουμε ετησίω ε, από 300.000 μάλλον θανάτους έχουμε ετησίω από αυτόν τον ε, βασικό λόγο, από αυτό το νόσημα και άλλα προβλήματα όπω την τύφλωση, ακροτεριασμού. Υπάρχουν οι εξή ε, λοιπόν δυνατότητε. Να πούμε ότι δεν είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Μια τέτοια πάθηση μπορεί να επιζήσει κανεί. Η δεύτερη επιλογή είναι να πούμε ότι η απουσία ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα αυτό είναι μέρο του προβλήματο και εγώ θεωρώ ότι πραγματικά απομένουν πολλά που πρέπει να κάνουμε και στον τομέα τη διάγνωση και τη περίθαλψη και στην επένδυση και στην έρευνα. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο το ψήφισμά μα ε, είναι επίκαιρο. Έχει ιδιαίτερη αξία και απεικονίζει τη συλλογική μα εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Ερχόμαστε τώρα στους υπολείπους ομιλητές. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Μάζε για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω το ψήφισμα αυτό και την προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας. Γνωρίζω εξαιδίας πείρας κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η προσέγγιση σας είναι πάρα πολύ θετική. Θα αυξηθεί οπωσδήποτε η συνειδητοποίηση του προβλήματος αυτό σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα δεν είναι μόνο η διαχείριση της νόσου αλλά και η πρόληψή της. Γιατί αυτό που έχει εδώ αποφασιστική σημασία είναι ακριβώς να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες περί τίνους πρόκειται, να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν εκ των προτέρων. Και επίση τι μπορούν να κάνουν ε, από τη στιγμή τη διάγνωση και μετά. Τι σημαίνει να αλλάξει τρόπο ζωή. Δεν σημαίνει απλώ ότι παίρνει φάρμακα, αλλά αλλάζει ακριβώ τον τρόπο που ζει. Και αυτό είναι ε, μια ευκαιρία για την κοινωνία των πολιτών, η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, να διαδραματίσει σημαντικό ε, ρόλο στην αύξηση της συνειδητοποίησης των πολιτών πάντα σε συνεργασία με τους ειδικού και εμπειρογνώμονες. Έχουμε λοιπόν εδώ μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε ε, συνέργειες και να συνεργαστούμε με όλους τους ενεχομένους στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Περέλο Ροντρίγκε για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε μια συγκυρία οικονομική κρίση και περικοπών στον προπολογισμό που επηρεάζουν τόσο τη δημόσια υγεία ε, όσο και γενικότερα, Στη δική μου περιφέρεια ε, δεν έχουμε ε, κονδύλια για την έρευνα. Σήμερα και αυτό ο, ο διάδοχος ε, της Ισπανίας, ο πρίγκιπας Φίλιππος. Θα πρέπει να αυξηθεί η έρευνα και στα βλαστικά κύτταρα θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα για τον τρόπο ζωής, τον τρόπο διατροφής. Γενικά θα πρέπει να βάλουμε την υγεία των ανθρώπων πρώτη προτεραιότητα και εκεί να γίνει έρευνα με εθνικά συντονισμένα προγράμματα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητάμε αποτελέσματα για το διαβήτη. Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων και όχι μόνο η ποιότητα και η ζωή τους η ίδια. Αυτοί που έχουν σήμερα προβλήματα τελικά θα είναι σε καλύτερη ζωή, καλύτερη ποιότητα ζωή και εμεί ω πολιτικοί θα έχουμε ανταποκριθεί στο καθήκον μα που είναι να φροντίζουμε και να προσέχουμε την υγεία των πολιτών. Αυτά τα ολίγα και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, η κυρία Μορκουνάιτε έχει ζητήσει το λόγο τώρα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. problema galima sakyti epidemija. skaičiai iš ties šokiruojantis 33 milijonai sergančių europos Sąjungos. Εδώ ξέρουμε ότι μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, δεκάδες εκατομμύρια, διατρέχουν κίνδυνο 300.000 θάνατοι ετησίων. Ο διαβήτη είναι ένα από τα πλέον Διορθώ, Διακόπτει ο Προεδρό. Συγγνώμη, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα ε, στη διερμηνία. Αν δεν σα πειράζει, θα σα παρακαλούσα να αρχίσετε ξανά την ομιλία σα από την αρχή. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα στο μεταξύ. Εδώ νομίζω συζητούμε ένα άκρο σημαντικό θέμα, γιατί το, το επιβεβαίωσε αυτό και η Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Είναι ε, μια από τι σοβαρότερε χρόνιε παθήσει παγκοσμίω ε, ο διαδίπη. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μια πραγματική επιδημία. Είπαμε ότι 32 εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο έχουν διαγνωστεί με διαβήτη. 10% του συνολικού πληθυσμού. Και άλλα 32 εκατομμύρια στη, βρίσκονται στην ομάδα κινδύνου. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο διαβήτη ασκεί μεγάλε πιέσει όχι μόνο στον τομέα τη υγεία αλλά και στη χρηματοδότηση της έρευνας, 10% ε, των δαπανών ε, του τομέα της οικονομικής περίθαλψης εκπροσωπεί διαβήτης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για να καταπολεμήσουμε αυτή την πάθηση και να στηρίξουμε την πρόληψη. Μόνο μισά, τα μισά από τα κατημέλη έχουν εθνικές στατικές κατά του διαβήτη. Και αυτό είναι από τα πρώτα βήματα στα οποία θα πρέπει να προβούμε. Η κοινωνία θα πρέπει να ασχοληθεί με το να εντοπίσει τους παράγοντες που προκαλούν το διαβήτη, τους παράγοντες κινδύνου. Θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικά προγράμματα και συντονισμένη δράση συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για την υγεία, για την ευαισθητοποίηση των θεμάτων υγεία, να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε ερευνά μα, να συμπεριλάβουμε εδώ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και πραγματικά εδώ θα πρέπει να συμφωνήσω με τον ε, κύριο Συγητή, τον κύριο Μπούζουτιλ, διότι πραγματικά θα μα δώσει τη σωστή πορεία για την καταπολέμηση αυτή τη ασθένεια στο ψήφισμα. Ευχαριστώ όλου του ομιλητέ και τι ομιλήτρε και ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye όπου ζητούν αυθόρμητα οι συνάδελφοι το λόγο. Ποιος θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό, παρακαλώ. Η κυρία Ζαπόρσκα πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το ψήφισμα απαιτεί συντονισμένη δράση των πολιτικών εθνών των κρατών μελών. Αναφέρονται βεβαίως και οι ευθύνε των πολιτών. Δεν έχουμε καμία εντολή βεβαίω να επιβάλλουμε την ανάληψη ευθυνών στους πολίτε. Από την άλλη όμως το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης θα έπρεπε να απηχεί τις ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσει για υγιή τρόπο ζωής. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα υγειονομική περίθελψης ε, να περάσει και στα χέρια των κρατών μελών. Στη Σλοβακία, λόγω χάρη, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η καταπολέμηση του διαβήτη με τρόπο γενναιόδωρο όπως σε χώρες πιο εύπορες. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η σωστή ενημέρωση για το διαβήτη στα διάφορα κράτη-μέλη. Η κυρία Γιούντιτ Μέρκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό και τους συναδέλφους. Σημαντικό το θέμα αυτό. Καλά που το φέρατε στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας για το εξή γεγονός. Όπως γνωρίζετε, το 1 τέταρτο των αρρώστων δεν το γνωρίζουν. Στην Ολλανδία είμαστε 16 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο διαβητικοί και το 1 τέταρτο το αγνοεί κιόλα. Ε, θα πρέπει να μάθουμε στον κόσμο τι να κάνει σπίτι του. Ε, έχει γίνει μεγάλη καινοτομία και χρειάζεται και μεγαλύτερη τεχνολογική πρόοδος για ένα smartphone, ας πούμε, να έχει ένα ημερολόγιο, να παρακολουθεί στο μητρό, ε, τι φάρμακα χρειάζεται ο καθένας και στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσουμε καλύτερα ε, για τέτοια ε, προγράμματα, να μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί τον εαυτό του και να κάνει και τη δοκιμή μόνος του για τη διάγνωση. Υπάρχουν λοιπόν ευκαιρίες για νέα υψηλή τεχνολογία και αυτό θα πρέπει να το έχουμε και στη στρατηγική, τη ψηφιακή ατζέντα για την ενεργό γύρανση. Θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε τέτοια προϊόντα και σε άλλες χώρες γιατί ε, χρειάζεται πραγματικά ελεύθερη κυκλοφορία της ιατρικής ε, και ενοτομίας. Μπορεί η περίθαλψη να είναι και πιο ευφυής και πιο τεχνολογική και ε, πιο σύγχρονη και να το μάθουν οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ακόμα ότι είναι ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούρσολ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εάν αναλύσουμε τα ποσά που αναφέρονται στην ε, επέκταση του διαβήτη τύπου Α ή Β στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε ξεκάθαρα ότι χρειάζονται σοβαρές προσπάθειες για την καταπολέμηση του διαβήτη και μάλιστα θα έλεγα την πρόληψη του διαβήτη. Σε αυτό επιμένω γιατί είναι και η πιο αποδοτική και σε οικονομικούς ακόμη όρους ε, λύση. Όταν μιλούμε όμως ε, για διαβήτη συνήθως ασχολούμαστε μάλλον με την θεραπεία παρά με την πρόληψη η οποία θα ήταν πολύ εύκολη με, μια, με έναν υγιεινό τρόπο ζωής θα μπορούσαμε να προλάβουμε την ε, πάθηση. Με, τον, ε, με το πρόγραμμα λοιπόν Ορίζον 2020 νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα, να έχουμε καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών προσπαθειών για το διαβήτη και να προ, βλέψουμε χρηματοδότηση των υποδομών. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόορη διάγνωση, για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. παπα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τον παιδικό διαβήτη, ένα θέμα που παρακολουθώ πολύ στενά και για ένα πρόσθετο προσωπικό λόγο, επειδή ενάμιση χρόνο πριν η εξάχρονη σήμερα νηψιά μου ένα μοναδικό παιδί διαγνώστηκε ότι πάσχει από διαβήτη τύπου α. θα θυμάμαι λοιπόν τις πρώτες προσπάθειες των γονιών θα θυμάμαι την προσπάθεια του πατέρα της να συνεννοηθεί με τον ασφαλιστικό του φορέα για να τους εξηγήσει ότι το ταμείο του έπρεπε να καλύπτει και τον ειδικό εξοπλισμό που χρειάζεται το παιδί για να μετράνε το ζάχαρο γιατί αυτό δεν είχε συμπεριληφθεί στις ρυθμίσεις που είχαν θα θυμάμαι ότι όταν το παιδί το πήγαν μετά τη διάγνωση στον παιδικό σταθμό που είχε γίνει δεκτό στο δημόσιο σταθμό και μετά από την καθοδήγηση και των γιατρών κάποιοι προσπάθησαν να πείσουν τους γονείς να πάνε πιο μετά το παιδί στο σχολείο για να μπορέσει όπως λέγανε να σταθεροποιηθεί. θέλω να πω δηλαδή για τα θέματα αυτά υπάρχει ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη ευρώπη μεγάλη άγνοια. υπάρχουν προκαταλήψεις υπάρχουν παρανοήσεις που τελικά οδηγούν και σε διακριτική μεταχείριση και αυτό όπως καλά γνωρίζω όλοι μας δεν το επιτρέπουμε και γι' αυτό ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρή και έντονη προσπάθεια γιατί και το παιδί που πάσχει από παιδικό διαβήτη θα μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά θα κάνει οικογένεια όπως όλα τα παιδιά θα ζήσει ευτυχισμένο όπως όλα τα παιδιά. σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η διάδοση της επιδημίας διαβήτη, η επέκταση της αποτελεί ένα από τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα της σύγχρονης ε, κοινωνίας. 90% όλων των παθήσεων ε, οφείλονται στον ε, διαβήτη τύπου Β που οφείλεται σε κακή διατροφή και ανεπαρκή φυσική άσκηση. Βλέπουμε τώρα ότι μετά τον ενήλικο πληθυσμό επεκτείνεται και στα παιδιά. Δυστυχώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Είναι όλο και πιο περίπλοκα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Πάσχων από διαβήτη σε όλη του τη ζωή. Και όταν γνωρίζουμε ότι με την βελτίωση των συνθήκων ε, ε, διατροφής και την ε, φυσική άσκηση θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό όταν ε, διαπιστώνουμε ότι θα μπορούσαμε παραδείγματι όπως έγινε με την αντιμετώπιση του καπνού με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και με προαγωγή φυσικών προϊόντων διατροφής ή ευαισθητοποίηση για τη φυσική άσκηση θα μπορούσαμε να αλλάξουμε την στάση των πολιτών και τη διάδοση του διαβήτη. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβει η Επιτροπή της Ευθύνες της και να εφαρμόσει αυτό το σύστημα, αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται στο κομμάτι ΚΑΤΣΤΙΑΙ με τον κύριο Νικολάτσικ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο διαβήτης εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 32 εκατομμύρια πολιτών ε, πάσχουν από διαβήτη και 325.000 θάνατοι καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του διαβήτη. Ο διαβήτης τύπου Β μπορεί να ε, μειώσει κατά 15 με, 20, κατά 5 με 10 χρόνια ζωής, το προσδόκιμο ζωής, ενώ ο τύπου Α έως και 20 χρόνια το κόστος ε, της θεραπείας του διαβήτη αντιστοιχεί στο 10% έως και 18,9% των συνολικών δαπανών ε, για την υγεία στα επιμέρους κράτη-μέλη. Χρειάζεται συντονισμός λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη υγεία νίκη στις αρμοδιότητες των ε, κρατών μελών θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα δράσεως για να προεγάγουμε ε, την υγιεινή διαβίωση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου να λάβουν το λόγο για να κάνουν τις ε, τελικές τους παρατηρήσεις ο κύριος Πίμπαλξ πρώτα. Πρόεδρε, νομίζω η κυρία Λούρφορτ και ο κύριος Παπα-Νικολαού ανέφεραν και το διαβήτη τύπου 1 και κάποια ζητήματα σχετίζονται και με αυτό το θέμα. Διότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ένα πρώτο θέμα, ώστε να ξεκινήσει η αγωγή όσο το δυνατόν συντομότερα. Το, το θέμα της έγκαιρης ε, διάγνωσης, λοιπόν, αυτό που ανέφερε ο κ. Παπα-Νικολάου, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε στη διαδικασία της περισυλλογής και των διαβουλεύσεων για τις χρόνιες παθήσεις εκπαίδευση των ε, γιατρών, των γενικών παθολόγων είναι και αυτό ένα στοιχείο, ώστε να υπάρχει διάγνωση έγκαιρη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζωτική σημασία. Για το διαβίτη τύπου 2 τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί η ευρωπαϊκή στατικική για τις, για τις χρόνιες μονοπαθήσεις όμως ε, υπάρχει η στατικική της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για τα θέματα παχυσαρκίας προβολικού βάρους, υγείας ε, και φυσικής άσκησης. Αυτή είναι εύστοχη στατικική. Σε συνδυασμό με τις εθνικές στατικικές στον τομέα αυτό θα μπορούσε να δώσει καρπούς. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή έχει πολλές διαστάσεις και θα συνεχίσει να τη για τη συζήτηση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καταπολέμηση του διαδίκτυου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Α, έχουμε ένα διαδικαστικό, παρακαλώ. Κυρία Λατφόρτ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να πω κάτι στον Επίτροπο. Νομίζω ότι δεν κατάλαβε αυτά που είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Άμα επιτρέπετε να μιλήσω εξ ονόματός του. Ε, μίλησε για το σχολείο του παιδιού. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τα γενικά θέματα των χρονιών νοσημάτων. Αν τα σχολεία είναι εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τι ειδικέ ανάγκε ενό διαβητικού παιδιού, κάνει ενέσεις ισουλίνη, μετράει το ζάχαρό του. Αυτά εννοούσε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Τι δουλειά έχουν τα χρόνια νοσήματα σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι παρανοήσατε πλήρω τι ειδικέ ανάγκε που έχει ένα διαβητικό, ιδιαίτερα τύπου 1 και όταν είναι παιδί. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Το κατάλαβα ότι ήταν διαβήτης τύπου 1, αλλά αυτό δεν αποκλείει ότι γενικώ θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση για την κατάσταση. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες, παρακαλώ η συζήτηση αυτή να λυθεί ε, και τώρα, εξ ονόματος του ε, Συμβουλίου, το λόγο έχει ο Υπουργό για να πληρώσει τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Ήταν σημαντική και καλή, κατά την άποψή μου. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να φέρουμε το διαβήτη στο επίκεντρο της προσοχής, όπως και τα άλλα χρόνια νοσήματα και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπουσουτήλ, την κυρία Λάτφορτ ε, και τους υπολείπους συντάκτες. για το γεγονός ότι ε, αναγνωρίζουν ε, τη στράτευση της Δανικής Προεδρίας στην προσπάθεια αυτή και ξέρετε ότι το τρίο της Προεδρίας ε, του Συμβουλίου ε, ασχολείται με αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας επιλέξαμε τα χρόνια νοσήματα, να ασχοληθούμε με αυτά, με ιδιαίτερο μοντέλο το διαβήτη, ως ιδιαίτερη προτεραιότητα. Η δική μου παρουσία σήμερα εδώ ξενόματος της Δανικής Κυβέρνησης εκφράζει άλλωστε αυτή την προσήλωσή μας. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας έδωσε να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις για τους πολλούς ανθρώπους που πραγματικά ε, ενέχονται σε αυτή την προσπάθεια και πάσχουν από την ασθένεια. Μαζί με τα κράτη-μέλη και ε, τους υπολοιπούς μπορούμε να δώσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στους διαβητικούς και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να αποφύγουν τα δεινά που περνούν σήμερα και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Γι' αυτό και για μένα είναι πολύ σημαντική η συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί, δεν σταματά εδώ, δεν τελειώνει σήμερα και θα ήθελα να σας υποσχεθώ ότι η Δανική Προεδρία μέχρι να ολοκληρωθεί το εξάμεινό της θα παραμείνει σε συνεργασία και με τις μελλοντικές προεδρίες για να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξη ε, της Ευρώπης αυτό το σημαντικό θέμα. Εύχομαι στο Κοινοβούλιο κάθε επιτυχία ε, στις επόμενες εργασίε, όπως και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω από κοινού να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα γιατί αφορά εκατομμύρια πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριε Προεδρεύον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σας και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και σα ενημερώνω ότι έχω λάβει τέσσερα ψηφίσματα για το θέμα αυτό Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι, ημέρα Τετάρτη. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 9 όπου και θα επαναληφθεί.